Αρχίζουμε τη συζήτηση δίνοντας το λόγο στον συντάκτη της ε, Συνδική έκθεσης, τον κύριο, την κυρία Μπόουλ. Με συγχωρείτε, κυρία Μπόουλ, για πέντε λεπτά. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, η προκάτοχός μου ως Πρόεδρος Οικονομικής και Νομισματικής Επιτροπής είχε καταθέσει να ψήφισμα στις 12 Μαρτίου του 2009. Από τότε δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα η άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σήμερα που είναι 8 Μαρτίου του 2009, εξακολουθούμε να περιμένουμε κάποια πρόοδο που ίσως θα επέλθει στις 8 Μαρτίου του 2011. Η Κομισιόν στην πρότασή της του Σεπτεμβρίου του 2009 εξέθεσε έξι τομείς προτεραιότητες και συμφωνούμε μαζί με αυτή την άποψη. Αλλά πάρα, πολλούς, πάρα πολλοί από αυτού που έλαβαν μέρο στη διαβούλευση που οργάνωσε η Κομισιόν είπαν ότι πρέπει να υπάρξει μια καταληκτική ημερομηνία για να υπάρχουν κίνητρα για αυτού οι οποίοι καθυστερούν να αποδεχτούν την πρόταση αυτή τη Κομισιόν. Δεν υπάρχει σαφέστερο τρόπο να το αναφέρουμε αυτό. Εμεί ζητούμε μια δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία να τεθεί μέχρι το αργότερο της 31 Δεκεμβρίου του 2020. Υπάρχουν όλο και περισσότερες αγορές και συμβάσεις που είναι διαμεθοριακού χαρακτήρα. Το να έχουμε κοινά πρότυπα για αυτές τις ε, πληρωμές, τις μεταφορές πιστώσεων κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την ανάπτυξη και την υγεία της ενέας αγοράς. Είναι πολύ καλύτερα για τους καταναλωτές να μην χρειάζεται να ελέγχουν αν υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις που ισχύουν στη μία χώρα ή σε μια άλλη ή να πληρώνουν κάποιο πρόσθετο κόστο λόγω αυτών των διαφορών. Επομένω, οι καταναλωτέ υποστηρίζουν αυτό το εγχείρημα. Πρέπει όμω να έχουν κάποια ασφάλεια και θα είναι πραγματικά ανησυχητικό αν δεν υπάρχουν οι απαραίτητε διασφαλίσεις για να μπορέσουν να ελέγχονται όλε αυτέ οι περιπτώσει των αμέσων πληρωμών. Ένα μεγάλο μέρο των <clears throat> εσόδων των τραπεζών προέρχονται από αυτές τις άμεσες συναλλαγές, αλλά δεν μπορούν να έχουν και την πίτα και τον σκυλοχορτάτο. Θα πρέπει να καταλάβουν οι τράπεζε ότι και οι καταναλωτέ αναρωτιούνται εάν είναι ασφαλή τα χρήματά του και αν κινδυνεύουν από αποτεώνε. Πολλά άτομα μπορεί να μην ε, προβαίνουν σε τέτοιε συναλλαγέ εάν δεν υπάρχει η απαραίτητη διασφάλιση. Θα πρέπει λοιπόν οι κατανοητέ να τύχουν των καταλληλών διασφαλίσεων. Δεν μπορεί κανείς να πιστεύει ότι οι τράπεζες θα βρουν όλες τις απάτες. Οι τράπεζες δεν τα κατάφεραν να αντιμετωπίσουν όλες τις περιπτώσεις με τις ε, ε, επιταγές και με τις απάτες οπισθογράφησης που οδηγούν στην καταβολή χρημάτων σε ένα λογαριασμό τρίτου. Αυτό μετά από πάρα πολλά χρόνια όταν κλείσανε αυτές τις τρύπε οι αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν είναι ικανοποιητικό λοιπόν με εμβαλωματικούς τρόπους και πρόσθετες υπηρεσίες να λύνονται αυτά τα προβλήματα, διότι έτσι δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια όλων. Δεν μπορούν να ληφθούν λοιπόν μέτρα απλώς μονάχα σε επίπεδο ε, κρά, κράτους μέλους, γιατί αυτά ευνοούν τις διαμεθοριακές απάτες. Όλα αυτά λοιπόν κύριε Επίτροπε θα πρέπει να τα λύσετε εσείς, να βρείτε τρόπους μέχρι τις 30, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2010 να κλείσετε όλες τις τρύπες που αφορούν τις άμεσες πληρωμές σε διαμεθοριακό χαρακτήρα. Είναι η κατάλληλη στιγμή λοιπόν να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή και να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν κάνει τα απαραίτητα σχέδια να συμμετάσχουν στις αρμόδιες έρευνες να το πράξουν. Τα κράτη-μέλη από μόνα τους δεν έχουν επιλύσει τα προβλήματα των εντολών για άμεσες πληρωμές. Θα πρέπει αυτά να προχωρήσουν σε άμεση λύση αυτών των προβλημάτων. Ίσως ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι τα ποσά τα οποία οι προμήθειες οι οποίες κρατώνται για πληρωμές με πιστοτικές ή χρεωστικές κάρτες. Και αυτό πρέπει να ληφθεί, με, το πρόβλημα με έναν τρόπο ο οποίος είναι συνάδων με την πολιτική ανταγωνισμού. Λέμε λοιπόν κύριε Επίτροπε, πρέπει επιτέλους να είσαστε στεναρός και να υπάρξει μια καταληκτική ημερομηνία ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι το σχέδιο αυτό για πληρωμές άμεσα σε όλη την ενιαία αγορά να πραγματοποιηθεί. Ευχαριστώ. Εξ ονόματος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρνιέ. Κύριε Μπαρνιέ, έχετε το λόγο. Ça marche. κυρίες και κύριοι βουλευτές, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. και θέλω να υποστηρίξω εξ αρχή αυτά που έλεγε προηγουμένω η κυρία Μπόλου. Λέγατε κύριε Μπόλου, ότι ο καταναλωτή χρειάζεται ασφάλεια. Συμφωνώ και σύμφωνα με μια φιλοδοξία που είχα πει για τη κράσεων στο Κοινοβούλιο να μπορέσει ο καταναλωτής να ανακτήσει την εσωτερική αγορά με συγκεκριμένα σχέδια. Αυτό περιλαμβάνει το σχέδιο του ενίου χώρου πληρωμών σε ευρώ του ΣΕΠΑ. Είναι ένα σύνθετο έργο. Αυτό που το, που το θέμα ωστόσο, απλές μεταφορές πιστώσεων στην Ευρώπη, δικαιολογεί τους στόχους μας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι, θα ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για την υποστήριξη που δίδει στο ΣΕΠΑ και για να απαντήσω στα πέντε ερωτήματα που θέσατε κύριε Πρόεδρε, που εντοπίζουν πολύ σωστά τα βασικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε. Θυμάμαι και την παλιά δουλειά και την εξαιρετικά θετική έκθεση και ενδιαφέρουσα έκθεση της κυρίας Μπερές και την έκθεση του κυρίου Γκοζές για, το, θέματα που, συν, που, ασχολούνται και τα, με το ΣΕΠΑ. Κυρία Πρόεδρε, έχουμε ένα ορόσημο. Ζητάτε μια τελική προθεσμία. Έχουμε μια τελική προθεσμία μια, θε, μια τελική δεσμευτική προθεσμία θα είχε πολλά θετικά. Σαφήνεια, προγραμματισμό επενδύσεων και πάυση συνύπαρξης δύο συστημάτων πληρωμών εθνικού και ευρωπαϊκού που δημιουργεί περιττό κόστος. Η δεσμευτική τελική προθεσμία θα προβλέπεται με νομοθετικό κείμενο. Εξετάζουμε πολλές εναλλακτικέ λύσεις. Πιστεύουμε του χρόνου το φθινόπωρο, το επόμενο ε, την επόμενη άνοιξη γνώμη θα έχουμε λήξει. Αυτή τη στιγμή είναι κάπως πρόημο να σας αναγγείλω μια συγκεκριμένη προθεσμία. Είδαμε την πρότασή σας για το 2012, θα το λάβουμε υπόψη, αλλά θα πρέπει να δώσουμε μια περίοδο προσαρμογής ε, για, τους, ε, για τις ε, τράπεζες, 12 ή 24 μήνες για τις μεταφορές και για τις εισφορές. Επίσης, άλλα θέματα που ασχολούνται, με τα οποία ασχολείται το ερώτημά σα. Πώς θα μπορέσει το ΣΕΠΑ να είναι χρήσιμο για τους χρήστες είναι κάτι που επίσης θα λύσουμε. Δεύτερο θέμα, ε, για την πολυμερή διαταμιπεζική προμήθεια. Είναι σημαντικό θέμα και για την εξέλιξη των καρτών και για την εξέλιξη των πληρωμών ΣΕΠΑ. Τέλη του 2009 η Κομισιόν ε, δημοσίευσε ένα κείμενο συζήτησης με νέα στοιχεία και με την άποψη των διαφόρων κατηγοριών χρηστών για το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε στα αποτελέσματα της δημόσιας αυτής διαβούλευσης. Το θέμα προφανώς ε, πρέπει να αναλυθεί και με το κατά πόσο είναι συμβατό με την ε, πολιτική ανταγωνισμού που είναι θέμα του συναδέλφου κ. Αλμούνια. Κάποιε παρατηρήσει ωστόσο μπορώ να κάνω. Για τι πληρωμέ για τις χρεώσεις. Μέχρι το 2012 θα υπάρχει δυνατότητα στην πολυμερή διαταπεζική προήθεια να καλύψει μέχρι 8 cents τις συναλλαγές, ε, τις συναλλαγές. Ωστόσο, 70% των ε, πληρωμών των χρεώσεων στην Ευρώπη γίνονται χωρίς καμία ε, πολυμερή διαταπεζική προμήθεια κάθε συναλλαγής. Η Επιτροπή λοιπόν η προμήθεια δεν θεωρείται ότι είναι ο μόνος μηχανισμός χρηματοδότησης, ούτε καν ο πιο αποτελεσματικός τέτοιος μηχανισμός. Για τις κάρτες, όπως ξέρετε η Επιτροπή ε, πήρε μια απόφαση κατά, κατά της διασυνοριακής προμήθειας στη Mastercard, το έκανε και για τη Visa. Για τη Mastercard η διαδικασία βρίσκεται σε έφεση στο ΔΕΚ. Ε, η συζήτηση αυτή αφορά το επίπεδο και τον τρόπο πλήρων καταβολή των προμηθειών αυτών. Το, η οριστική απόφαση του ΔΕΚ θα συμβάλλει σε μια καλύτερη νομική ασφάλεια. Τρίτο θέμα. Είχα την ευκαιρία να το πω και στην ακρόασή μου. Είμαι υπέρ του να ξεκινήσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στον τομέα των καρτών μια σειρά πρωτοβουλειών συζητώνται αυτή τη στιγμή στον ιδιωτικό τομέα, Money, Payfair και άλλα. Θα συναντηθώ κυρία Πρόεδρε και κυρίες βουλευτές με τους φορείς της αγοράς για να εξετάσω από κοινού την δυνατότητα να προχωρήσουμε και να συντονίζουμε τις ε, πρωτοβουλίες ε, στο πλαίσιο ευρύτερη δράσης. Επιπλέον η Επιτροπή θα αναλύσει με βάση τους κανόνες ανταγωνισμού τα επιχειρήματα που παρουσιάζουν τα συστήματα κρατών για να δικαιολογούν τον τρόπο χρηματοδότησή τους. Τέταρτο σημείο. Σε ό,τι αφορά το μέλλον της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης ε, και της διαχείριση, ξέρετε, δεν θέλουμε μια πανευρωπαϊκή διαχείριση. Γι' αυτό υπάρχει κοινή ε, δημιουργία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για να δημιουργηθεί ένα συμβούλιο ΕΠΑ που θα έχει μικρό αριθμό εκπροσώπων υψηλού επίπεδου από τον κλάδο και τους χρήστες που θα διευκολύνει το, τον διάλογο και θα επιτρέψει μια καλύτερη αντιμετώπιση της κατάστασης. Η πρώτη συζήτηση θα γίνει την Άνοιξη και είναι προφανές κυρίες και κύριοι ότι προσωπικά θα ενημερώνω το Κοινοβούλιο προσεκτικά και στενά για τις, ε, διαδικασίες, για τις εργασίες στο Συμβούλιο ΣΕΠΑ όταν συζητήσουμε ιδίως στην Επιτροπή Οικονομικών Οικονομική πολιτική. Τελευταίο θέμα. Πώ λαμβάνονται υπόψη τα, συμφέροντα των τελικών χρηστών. Κύριε Πρόεδρε, εγώ λυπούμε που ο κλάδο ε, συχνά ε, φαίνεται ότι είναι επιφυλακτικό και δεν θέλει να λάβει υπόψη τι ανησυχίε των καταναλωτών. Υπάρχουν πιθανές Βελτιώσει στην διαχείριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών για την διευκόλυνση της διαφάνειας και την λήψη υπόψη των χρηστών. Το Συμβούλιο ΣΕΠΑ θα αποτελεί μια καλή πλατφόρμα για τι βελτιώσει βελτιώσεις αυτές. Έχω επίσης την πρόθεση να αναλάβω δράση σε συγκεκριμένα ζητήματα, ιδίω τι βελτιώσει που πρέπει να επιφέρουμε στα συστήματα χρέωση η Επιτροπή και η Κεντρική Τράπεζα θα στείλουν ε, μια επιστολή στο Ευρωπαϊκό Συμβείο Πληρωμών ζητώντας να συμπεριλάβουν κάποιες αλλαγές που θα καλύπτουν την ανάγκη, τις ανάγκες των καταναλωτών. Δεν αποκλείω η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν εμπόδια στο δρόμο αυτό για να καλυφθούν ακριβώς οι ανάγκες των καταναλωτών. Όπως θα καταλάβατε κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είμαι αποφασισμένος να δράσω και να επιτρέψω την λειτουργία, τη σωστή λειτουργία του ΣΕΠ, όπως σας το είπα τον Ιανουάριο, θα ε, προσπαθήσω να βελτιώσω την κατάσταση μέσω και της ε, κοινοβουλευτικής δραστηριότητα και του ψηφίσματος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο. Εξ των πολιτικών ομάδων, πρώτο ο κύριος Γκουζές για δύο λεπτά. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δεν αμφιβάλλω για την αποφασιστικότητά σας και με τα στοιχεία που μας δώσατε ήδη δώσατε μια απάντηση στις περισσότερες ερωτήσεις που είχαμε. Ερωτήσεις που τίθενται από το ψήφισμα αυτό. Απλώ θέλω να πω ότι η δυσκολία του θέματο ε, συνίσταται στο ότι το ΣΕΠΑ είναι μια πρωτοβουλία των πιστοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων των τραπεζικών κυρίω ιδρυμάτων και η οδηγία για τι υπηρεσίε πληρωμών ε, που ήμουν εγώ εισηγητή για το θέμα αυτό είχε ω αντικείμενο να μα επιτρέψει να μπορέσουμε να καθορίσουμε τα απαραίτητα νομικά μέσα για να δημιουργήσουμε αυτό το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληρωμών. Επίσης, είχε ως αντικείμενο να βελτιώσει τον ανταγωνισμό στον τομέα των πληρωμών και ο τίτλος 2 προβλέπει τη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών ε, που θα έσπαγαν το μονοπόλιο των τραπεζών. Ε, αυτή η διαδικασία λοιπόν εξηγεί ένα μέρος της καθυστέρησης. Είναι αλήθεια όμως, όπως είπατε κι εσείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα τραπεζικά ιδρύματα έδειξαν απροθυμία στην εφαρμογή αυτών των μέτρων και υπάρχει μια εξήγηση, δηλαδή το κόστος. Και για να σας δώσω μια ιδέα για το κόστος, πράγμα το οποίο θα γνωρίζετε, στη Γαλλία το κόστος για την εφαρμογή του ΣΕΠΑ είναι ίσο και υψηλότερο από ότι το κόστος του περάσματος στο ευρώ. Υπήρξε και το θέμα της Επιτροπής Συναλλαγών που πρέπει να το εξετάσουμε έχοντας κατά δύο θέματα. Πρώτον, όπως υπενθυμίσετε και είναι το θέμα της συμβατότητας με τους κανόνες του ανταγωνισμού και δεύτερον, το δεύτερο στοιχείο που δεν πρέπει να μελήσουμε είναι ότι οι υπηρεσίες πληρωμών είναι μια εμπορική δραστηριότητα των Ιδρυμάτων Πληρωμών και γι' αυτό πρέπει να ανταμείβεται επαρκώς και δεν θέλαμε να υπάρχει μια δυνατότητα μονομερούς αφαίρετης μονομερούς καθορισμού διατραπεζικών ορίων κέρδους που θα ήταν υπερβολικά. Κύριε Πέτροπε, λοιπόν, εμεί ε, βασιζόμαστε σε εσά, ούτω ώστε αυτή η πρόοδο για τη δημιουργία τη ενιαία αγορά πληρωμών σύντομα να μετατραπεί σε δημιουργία ευρωπαϊκών οργάνων ε, μεταφορών και μεταφορά πιστώσεων. Ευχαριστώ ο Ευρωπαϊκός, ο ενιαίος χώρος πληρωμών ευρώ είναι ένα σημαντικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Και είπε και ο συνάδελφος κύριος Γκοζές ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι προτάθηκε και η πολιτική μας ομάδα το υποστηρίζει πλήρως και προσωπικά δεν ε, διαφωνώ καθόλου να τεθεί μια ε, τελική προθεσμία για την εφαρμογή που θα μπορούσε να ε, μην εξαρτάται από του 3, 4 ή 5 μήνε για τη σωστή λειτουργία του συστήματο. Μα ενδιαφέρει να λειτουργεί όμω σωστά το σύστημα. Και για να λειτουργεί σωστά, και αυτό αποτελεί και μια έκκληση προ τον κλάδο, πρέπει να είναι φιλικό το σύστημα αυτό προ το χρήστη. Δεν θέλουμε να υπάρχει κάποια κρυφή αντίσταση. Δεν θέλουμε ε, να υπάρχει δυσπιστία ε, έναντι του συστήματος. Θέλουμε ε, το σύστημα αυτό να είναι φιλικό προς αυτούς που θέλουν να το χρησιμοποιήσουν πραγματικά. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Και το δεύτερο θα πρέπει να είναι κάτι που θα βοηθά τη λειτουργία της οικονομίας. Και αυτό ε, ισχύει και για το σύστημα υπολογισμού ε, της άμεσης χρέωσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ένα λογικό μοντέλο το οποίο μπορώ αυτή τη στιγμή να σας προτείνω. Θα πρέπει η ίδια η οικονομία να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και να παρουσιάσει, να προτείνει ένα τέτοιο νέο μοντέλο που να λειτουργεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν, κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως λέει και αυτό το σχέδιο ψηφίσματος, μέσα σε μια δεδομένη προθεσμία, μέσα στο 2010, να υποβάλει μια συγκεκριμένη πρόταση, διότι δεν μπορούμε μπορούμε να αφήσουμε ε, χωρίς τελική προθεσμία αυτή την ε, πρωτοβουλία. Είναι μια πρωτοβουλία που ε, θα πρέπει να συνεχιστεί με πρακτικά βήματα και χρειάζεται μια κοινή πρωτοβουλία για να λειτουργήσει αυτό συνολικά. Αυτή είναι η δική μας πρόταση για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ähm, είναι θετικό το ότι έχουμε το ευρώ. Ε, το χρειάζονται οι μικρές χώρες και η δική μου χώρα, η Αυστρία, ε, τέθηκε υποπίεση το 2007 με την ε, οικονομική κρίση και καταλαβαίνουμε τη σημασία που έχει. Από την άλλη πλευρά καταλαβαίνουμε τις συνέπειες και τις ε, ε, αρμοδιότητες που υπάρχουν και γι' αυτό ρωτώ την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποιος είναι υπεύθυνο για την κρίση στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ποιος είναι υπεύθυνο γιατί έφτασαν ασφαλμένα στοιχεία από τον προπολογισμό από την Ελλάδα και τρίτον δεν είναι πραγματικά η Ελλάδα το πρόβλημα όπως είναι η Ισπανία το πρόβλημα και τέταρτον μπορούμε, μπορεί να εγγυηθεί η Επιτροπή ότι δεν θα υπάρξουν ασφαλμένα συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα υποβάλλονται για του προπολογισμού, τι κάνει από αυτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και θα πρέπει τελικά αυτοί οι οποίοι έχουν την ευθύνη να είναι τελικά υπόλογοι και να ζητηθούν ευθύνε. Μπορούμε να εγγυηθούμε ότι επιτέλους θα τηρούνται οι κανόνες του παιχνιδιού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέρμπερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι σημαντικό το ότι μιλάμε για, ε, ένα, για μια ενιαία διαδικασία που θα ανταποκρίνεται σε ένα ενιαίο νόμισμα και νομίζω ότι είναι σωστό να έχουμε κατά νου μια ενιαία διαδικασία ε, σε ένα ενιαίο ε, χώρο πληρωμών. Κάτι τέτοιο πρέπει να λειτουργήσει και θα πρέπει αντίστοιχα να προσαρμοστούν και οι κανονιστικές διατάξεις. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα που το σύστημα άμεσης χρέωσης ε, είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο και ε, είναι ένα σύστημα το οποίο απλουστεύει τη διαδικασία το σύστημα το οποίο προτείνεται ε, ω κανονιστικό σύστημα είναι γραφειοκρατικό και πολύπλοκο και γι' αυτό θα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο κύριε Επίτροπε αν ε, μπορεί να μπει μια τελική προθεσμία ε, μέσα στην οποία πρέπει να επανεξεταστεί αυτό το σύστημα και θα πρέπει να υπολογίζονται τα τέλη χρεώσεων ούτω ώστε να οδηγήσει το σύστημα σε μια λογική και απλή διαδικασία στην οποία να μπορούν να βασίζονται οι επιχειρήσει. Και Γι' αυτό συμφωνώ με αυτή την πρόταση ψηφίσματος και θα πρέπει η διαδικασία στα κατι μελη να αξιολογηθεί και μετά την τελική εισαγωγή αυτού του συστήματος ε, του ενιαίου χώρου σε ευρώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάρας για δύο λεπτά. Κύριε Επίτροπε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σχετικά με τις απαντήσεις του Επιτρόπου στην προφορική ερώτηση. Θεωρούμε ότι είναι σωστές οι απαντήσεις του και τον ευχαριστούμε. Ανταποκρίνονται στους στόχους που έχει θέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι ότι η μέθοδος ε, της αυτορύθμισης που είχαμε επιλέξει μέχρι τώρα στον ε, τραπεζικό τομέα όπου θέλουμε εκατοντάδες τράπεζες ε, να ενταχθούν σε αυτό το σύστημα ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ως τμήμα της ενιαίας αγοράς. Ο χώρος ΣΕΠΑ είναι μεγαλύτερος από το χώρο του ευρώ και εγώ είμαι υπέρ ενός ενιαίου συστήματος ε, για τον υπολογισμό των δεδομένων για να ρυθμιστούν τα ανοιχτά ζητήματα και να είναι νομικά δεσμευτικό το σύστημα. ούτως ώστε ο χώρο ΣΕΠΑ το συντομότερο δυνατόν και όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά να τεθεί σε λειτουργία. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, όντως η ΣΕΠΑ είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία η οποία οπωσδήποτε θα ωφελήσει καθώς επίσης και θα βελτιώσει την παρούσα κατάσταση όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές ε, πληρωμές και θα δημιουργήσει μια ενιαία αγορά πληρωμών πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορεί κανείς όπου και αν βρίσκεται ή όπου και αν χρησιμοποιεί αυτού του ίδιου στις ε, υπηρεσίες να μπορεί να προσφύγει σε αυτό το ενιαίο μέσο εργαλείο πληρωμών. Επίσης ε, θα ε, μειωθεί το κόστος μετακίνησης κεφαλαίων από περιφέρεια σε περιφέρεια που υπολογίζεται περίπου ε, στο 3% του ΑΕΠ. Θα θυμάστε ότι ο ίστατος στόχος της ΣΕΠΑ ήταν ακριβώς να δημιουργήσει ένα βιώσιμο εργαλείο ε, για ολόκληρη την ε, Ευρώπη και βεβαίως αυτός ο τόσο φιλόδοξος στόχος είναι ε, δύσκολος κυρίως την στιγμή που χρειάζεται κανείς να βρει και κάποιες συμβαστικέ λύσεις έτσι ώστε να ικανοποιηθούν τα αντικρουόμενα αιτήματα Τη της ε, πανευρωπαϊκής ε, τραπεζικής αγοράς. Ε, κυρίως δεν λαμβάνοντας υπόψη και την πρόσφατη κρίση, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα. Νομίζω ότι θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις, θα πρέπει ε, να ε, εκπονηθεί ένα λογικό ε, και θεμητό χρονοδιάγραμμα. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Κάρας προηγουμένως. Επίσης η έννοια ότι εγχώριες αρχές θα μπορούν να ισχύσουν ταυτόχρονα με τη ΣΕΠΑ θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και σίγουρα δεν θα βοηθήσει την πραγματική εφαρμογή της ΣΕΠΑ. Θα πρέπει οπωσδήποτε να να ε, υπάρξουν δεσμευτικές αρχές όσον αφορά την μεταπίδηση στις αρχές ΣΕΠΑ. Η κυρία Μπασέσκου για ένα λεπτό. Κύριε eh, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας πω ότι η χώρα μας ε, θέλει να προσχωρήσει σε αυτό το φορέα και το 2009, το 2007. Το 2009 μεταφέρθηκε στην ιστορικομαστική και αυτή το 2007 και μετά η Ένωση Τραπεζών ε, έχουμε αναλάβει τις αναγκαίες ενέργειες ούτως ώστε να μπορεί να μπει στη ΣΕΠΑ η χώρα μας. Οπότε τώρα έχουμε προχωρήσει σε αυτό το σύστημα του, των πληρωμών και ορισμένες τράπεζες επίσης μπορούν να κάνουν άμεση χρέωση τα μέσα επόμενα χρόνια. Επομένως, η πρόοδος που σημειώνουμε είναι αναμφίβολη και οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΤΕ, οι, οι ασφάλειες θα μπορούσαν να έχουν κάνει ό,τι χρειάζεται ώστε να μπορούσαν να προσχωρήσουμε στον ενίο αυτό χώρο και όλος ο κρατικός τομέας μόλις μπορούμε να μπούμε και στο ευρώ. Νόμος της Επιτροπής, ο κύριος Μπαρνιέ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω έναν έναν όσους πήραν το λόγο για να πούν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και μετά και από την αρχική τοποθέτηση της κυρίας Σάρον Μπόουλς βλέπω ότι υπάρχει ομόθυμη αντιμετώπιση του θέματος ε, από την Ολομέλεια. Ο ενιαίος χώρος δεν αφορά μονάχα και συγκεκριμένα τις ε, πληρωμές, ε, αφορά ένα πολύ γενικότερο πρόγραμμα και πραγματικά ε, με μεγάλη ικανοποίηση ακούω την συνένεση η οποία εκδηλώνεται από πλευρά του Κοινοβουλίου και βλέπω ότι όλοι επιθυμούν να θεσπιστεί δεσμευτική ημερομηνία. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα μικρό περιθώριο χρόνου έτσι ώστε να υπάρξει μια διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους. Η διαβούλευση αυτή θα είναι ταχεία ε, και ε, ε, πραγματικά όσον αφορά την εφαρμογή της ΣΕΠΑ θα λάβω τις αποφάσεις μου σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι η ΣΕΠΑ ε, μπορεί να δώσει θετική απάντηση στα μελήματα των ε, μικρών επιχειρήσεων, ε, στα, στις των επιχειρηματιών, αλλά και γενικότερα όλων των εμπλεκομένων μέρων. Καταλαβαίνουμε ότι ε, θα ήταν πάρα πολύ καλό και προς το συνολικό συμφέρον ε, να ε, διευρυνθεί η ΣΕΠΑ. Ξέρω ότι ήδη στη χώρα σας ισχύει και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα είναι δεσμευτική για όλους. Όπως είπα και προηγουμένως, θα έρθω σε επαφή με τους εμπλεκόμενους φορείς. Θα κάνω όσο γίνεται πιο γρήγορα την διαβούλευση έτσι ώστε ε, να δούμε τα διάφορα επιμέρους ζητήματα όπως ας πούμε την ενδεχόμενη μελλοντική χρηματοδότηση ενός ε, μοντέλου πανευρωπαϊκής ε, κάρτας καθώς επίσης ε, και ε, όλων των ε, επιμέρους ζητημάτων που αναφερθήκατε και εσείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπατε που ευθυγραμμίζονται με τις ανησυχίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Όλους τον κύριο Επίτροπο, όλους τους ομιλητές, έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος ως περάτωση αυτής της συζήτησης εξ ονόματος Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Η συζήτηση έληξε, ψηφοφορία Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Το επόμενο σημείο της της διάταξης είναι η έκθεση του κυρίου Λένε σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς εταιριών ορισμένων μορφών όσον αφορά τις μικρομονάδες. Ο κύριος Λένε, ο εισηγητής, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην έκθεση αυτή πρόκειται για